Ηρακλήδη, τονίζω και πάλι ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στα εξωτερικά μα σύνολα είναι κάτι που μα ανησυχεί. Θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τους γειτονέ μα και τα διεθνή δεσμικά όργανα. Ε, επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσου συνεργαστήκαμε στο ανθρωπιστικό μέτωπο. Θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης να βοηθήσει ούτως ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση εξωτερικά σύνορα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, Ευχαριστούμε Υπουργέ και τώρα εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επίτροπο Ντάλι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Υπουργέ, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. Σα ευχαριστώ για αυτή τη σημαντική συζήτηση. Η ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα που μας ανησυχεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τον συμβασμό των δικαιωμάτων των προσφύγων, των ετούντων άσυλο και των μεταναστών τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη γειτονία μας. Κάθε μορφή βίας εναντίον προσφύγων και μεταναστών δεν χρειάζεται βεβαίως να το πω, είναι απαράδεκτη. Ο σεβασμός στα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου θα πρέπει να εξασφαλίζεται χωρίς καμία εξαίρεση. Τα κράτη-μέλη πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με αυτές τις αρχές όταν εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων, το άσυλο και τις επιστροφές. Δεν επιτρέπονται οι αποθήσεις. Η πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου και ο σεβασμός στην ε, αρχή και η μη επαναπροώθηση πρέπει πάντοτε να εξασφαλίζονται. Τα κράτη-μέλη έχουν ε, θεσπίσει μηχανισμούς για την αποφυγή των ε, επαναπροωθήσεων. Πρέπει επίσης όμως να εξασφαλίσουν ότι θα έχουν δομές και μηχανισμούς ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα στις προκλήσεις. Οι προκλήσεις στα εξωτερικά μας σύνορα είναι πολλές και η Κομισιόν βρίσκεται σε διαρκή και μόνιμη επαφή με τα κράτη-μέλη και τους παρέχει βοήθεια συμπεριλαμβανομένης και ε, εκπαίδευσης ε, για τους σύνοροφύλακες ώστε να ε, δρούν ε, με βάση το πνεύμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επίση, η Κομισιόν παρακολουθεί στενά την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα και βρίσκεται συνεχώ σε επαφή με τα κράτη-μέλη όσον αφορά τι κατηγορίε μη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο στα ε, εξωτερικά σύνορα. Ω θεματοφύλακα τη συνθήκη, η Κομισιόν θα αναλάβει κάθε απαραίτητη δράση όπου αυτό κρυθεί αναγκαίο. Επίση, έχουμε πλέον ένα νέο Frontex που έχει ενισχυμένη εντολή και με ακόμα μεγαλύτερη επικέντρωση στην ανάγκη να γίνονται σεβαστά τα θεδομελιώδη δικαιώματα. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, συντάχθηκε και η νέα στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα από την ίδια την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Διορίστηκε και αξιωματούχος θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο οποίος συμβάλλει στην εφαρμογή των θυμολογικών δικαιωμάτων από τον οργανισμό και παρακολουθεί την κατάσταση. Αυτός ο μηχανισμός θα αξιολογεί την ε, συμμόρφωση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του Frontex σε όλες τις δράσεις του. Θα είναι τα αυτιά και τα μάτια του αξιωματούχου ε, δικαιωμάτων. 40 τέτοιους ελεκτές πρόκειται να προσλάβει ο Frontex έως τις 5 Δεκεμβρίου του 2020. Επίσης, έχει δημιουργηθεί ένας ε, μηχανισμός υποβολής παραπώνων που επιτρέπει σε όλα τα άτομα που εμπλέκονται ή πλήττονται από δράσεις ε, του οργανισμού ε, ή που με τον οποιοδήποτε τρόπο έχει έρθει σε επαφή με αυτόν τον οργανισμό που θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά του να υποβάλει τέτοια καταγγελία γραπτός στον ίδιο τον οργανισμό. Το, αυτά που συμβαίνουν στα εξωτερικά μας σύνορα επηρεάζουν την Ευρώπη. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε υποστήριζε τους εταίρους μας στα εξωτερικά σύνορα και τους πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στις χώρες αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί παγκόσμιο παίκτη όσον αφορά την ε, παροχή βοήθεια σε πρόσφυγες και μετανάστες, ιδίως σε γειτονικές χώρες και όσον αφορά την υποστήριξη των γειτονικών χωρών ε, στην, όσον αφορά την ικανότητά τους να αντιμετωπίζεται η λαθροδιακίνηση ανθρώπων. Για παράδειγμα, υποστηρίζουμε την Τουρκία που φιλοξενεί πάνω από 4 εκατομμύρια μετανάστες. Έχουν κινητοποιηθεί πλήρως τα 6 δισεκατομμύρια του μηχανισμού και έχουν αποφέρει πραγματικά απτά αποτελέσματα. Πάνω από 1,7 εκατομμύρια πρόσφυγες ωφελούνται από το Δίκτυο ασφαλείας έκτακτης ανάγκης που είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ανθρωπιστικό πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί ποτέ. Επίσης υποστηρίζουμε πάνω από 500.000 πρόσφυγες παιδιά να πάνε στο σχολείο. Θέλουμε οι συνοριακές αρχές να είναι αξιόπιστο εταίρος για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ωστόσο, οι ικανότητε υποδοχής, ιδίω στη Σερβία και την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, έχουν εξαντληθεί. Και πολλές φορές οι μετανάστες βρίσκονται και ζουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Χρειάζεται περισσότερη βοήθεια, οικοδόμηση ικανοτήτων, ώστε οι χώρε αυτέ να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην ανάγκη να διαχειρίζονται την μετανάστευση, να αντιμετωπίσουν τις δευτερογενείς ε, μετακινήσεις, αλλά με ταυτόχρονη ανθρώπινη μεταχείριση των προσφύγων και των μεταναστών. Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει τεχνική βοήθεια μέσω των προγραμμάτων ε, προενταξιακής βοήθειας στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν τα εθνικά συστήματα διαχείρισης μετανάστευσης. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα παρέσχε 135 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετη βοήθεια στη Σερβία, την Βόρεια Μακεδονία και την Βοσνία Ερζεγοβίνη μέσω του ε, εργαλείου για την προενταξιακή βοήθεια και 32,6 εκατομμύρια ευρώ μέσω τη Ευρωπαϊκή Ανθρωπιστική βοήθεια. Σε όλε αυτέ τι δράσει, εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, η προστασία των πλέον ευάλωτων, ιδίω των παιδιών και των ασυνόδευτων ανηλίκων, παραμένουν ύψιστη προτεραιότητα για την Κομισιόν. Η Κομισιόν κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να βοηθά τα κράτη-μέλη ώστε να αντιμετωπίσουν την κατάσταση στα εξωτερικά μας σύνορα. Η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων ατόμων πρέπει να εξασφαλίζεται και να προστατεύεται. Πολλά έχουμε επιτύχει. Όμως χρειάζεται να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια κοινή αντίληψη για το πώς συλλογικά θα διαμορφώσουμε και θα διαχειριστούμε τις πραγματικότητες που δημιουργεί η μετανάσταση. Πρέπει να ενωθούμε γύρω από τις κοινέ μας αξίες και τις ανθρωπιστικές μας ευθύνες και να προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο ολοκληρωμένη, πιο ενιαία ε, την, ε, τις κοινωνίες της Ευρώπης. Βασίζομαι στη δική σας υποστήριξη καθώς και στην υποστήριξη του Συμβουλίου. Ευχαριστούμε Άφνα, ευχαριστούμε Επίτροπε και τώρα ξεκινάμε με τις παρεμβάσεις εκ των πολιτικών ομάδων. Προφανώς ξεκινάμε με το ΕΛΚ. Ο κύριος Ράντεφ, για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ συνάδελφε. Ευχαριστώ συνάδελ, πρόεδρε, συνάδελφοι. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο δρόμος των Δυτικών Παλκανίων είναι ο βασικότερος δρόμος πρόσβασης στην Ευρώπη. Και είναι και ένας από τους πιο πολυσύχναστους. Δυστυχώ, τα κράτη-μέλη που βρίσκονται πιο κοντά, η Κροατία, η Ελλάδα και ούτω καθεξής, πρέπει να φορτωθούν ένα ε, δυσανάλογο μερίδιο ευθύνη λόγω τη γεωγραφικής εγκύτητας. Βλέπουμε τι συμβαίνει στα σύνορα μεταξύ Κροατίας και Βοσνίας Ερζεγοβίνης και επίσης βλέπουμε τι συμβαίνει και στα ελληνικά νησιά. Δεν σταματάνε να φτάνουν φάρκες και σκάφη με μετανάστες. Ε, δεν ζητούν διεθνή προστασία μόνο στα επίσημα ε, σημεία ελέγχου. Κοιτούν να περάσουν τα σύνορα σε σημεία που δεν ελέγχονται. Και επίσης υπάρχουν και τα δίκτυα των λαθρεμπόρων, οι οποίοι προσπαθούν να προωθήσουν τους μετανάστες προς τη Δυτική Ευρώπη το 2018 λόγω της υψηλής μεταναστευτικής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έδωσε 2,6 εκατομμύρια στην ε, Κροατία για να βελτιώσει την ε, προστασία των εξωτερικών συνόρων. Αυτό έγινε βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων ώστε τα μέτρα που λαμβάνονται στα εξωτερικά σύνορα να είναι αναλογικά να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα και να μην υπάρχει παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου στον τομέα του ασύλου. Στι αρχέ του 2018, 36 εκατομμύρια ευρώ ε, απεστάλησαν στην Βοσνία Ζεγοβίνη, ακριβώ για να ε, φροντίσει τι κατεπίγουσε ανάγκε μεταναστών και προσφύγων εκεί. Δεν προστατεύουμε απλώ τα εξωτερικά μα σύνορα, διότι εάν γίνεται σεβαστό ο νόμο, η νομοθεσία και οι διεθνεί συμβάσει, πρέπει να σεβαστούμε και τα θεμελιώδη δικαιώματα και την εξωπρέπεια των μεταναστών. Η Κροατία και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προστατεύουν δεόντω τα εξωτερικά μα σύνορα και κάνουν ό,τι μπορούν για του κανόνε. Ευχαριστώ να τηρείτε το χρόνο ομιλία, αν γίνεται. Ε, και τώρα, εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο λόγο στην κυρία Πύρη για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ κάτι. unprecedented peak in refugee arrivals in 2015 το 2015 είχε φανεί το ότι έχουμε κενά στην ε, πολιτική μας ε, και είχαμε πέντε χρόνια από τότε για να βρούμε λύσεις. Όμως, σε πολλά σημεία η κατάσταση στα συνοραντή να βελτιωθεί, επιδεινώνεται. Συνεχώς. Βλέπουμε άπραγοι εγγύους να χάνουν τη ζωή τους στην ε, Μεσόγειο. Χιλιάδες ζουν σε στρατόπεδα και ασυνόδευτοι ανήλικοι, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ασύλου πολλοί αναγκάζονται να γυρίσουν σε χώρες μη ασφαλείς. Ε, στα κέντρα κράτησης έχουμε τις επαναπροωθήσεις. Αυτά δεν είναι λύσεις. Ελπίζουμε ότι η Προεδρία θα λάβει υπόψη τα όσα λέμε εδώ ε, και αυτά θα ζητούν στο Συμβουλίο. Ας μην ξεχνούμε ότι οι χώρες της Μεσογείου αναδέχονται τους περισσότερους πρόσφυγες, αλλά επίσης κάποιοι ε, ε, γειτονές μας και αυτοί δεν κάνουν ε, τίποτα. Θα πρέπει τι γίνεται με Μαρόκο και Τουρκία. Πολλές φορές εδώ μιλούμε για ευρωπαϊκές αξίες και χρειάζεται σεβασμός αξιοπρέπειας και δικαιωμάτων. Αυτό ισχύει και για τους πρόσφυγες που ζητούν την προστασία και σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και τώρα για το Renew Europe ο κύριος Ασμάνη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο που ήρθαν απόψε. Ήρθε η ώρα να απεμπλακεί η κατάσταση στο μεταναστευτικό. Αυτό το οφείλουμε στους συμπολίτε μας. Θα πρέπει να βρούμε μια λύση να μας κάνει πρωτοπόρους. Κάτι να γίνει και με την περιοχή ε, Σέγγεν και με τα εξωτερικά σύνορα. Έχουμε το νέο σύμφωνο και το Renew έχει μια προσέγγιση σφαιρική. Το προτείναμε ως δέσμη μέτρων την περσμένη εβδομάδα για να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε την πίεση στα σύνορά μας. Χρειάζονται νέες συνεργασίες με τις τρίτες χώρες στο μεταναστευτικό. Είναι αυτός ο μόνος τρόπος. Εν τω μεταξύ χρειάζεται μια κοινή προσέγγιση για όσους φτάνουν παράνομα. Χρειάζεται καταγραφή, άματη αφήξη και έλεγχη ασφαλείας. Ανθρωπίνες συνθήκες υποδοχής και να μπορούμε να κάνουμε έναν υπολογισμό το ποιοι θα τύχουν ασύλου και ποιοι όχι. Να δούμε όλοι μαζί σαν κοινή υπευθυνότητα ποιοι χρήζουν προστασίας, ποιοι πρέπει να επιστρέψουν σε χώρες που είναι ασφαλείς. Για αυτό το νέο πακέτο έχουμε υψηλές προσδοκίες. Και ελπίζουμε και το Συμβούλιο να συμφωνήσει, αλλά για πέστε μας, συμφωνείτε με το Renew Europe ότι θα πρέπει να αναβαθμίσετε τις προσπάθειές σας όταν κάποιο κράτος μέλος εξωτερικά σύνολα δεν θέλει ή δεν μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει γιατί αυτό έγινε στο παρελθόν. Τι θα κάνει η Κομισιόν για τις ροές των μεταναστών στο εσωτερικό της Ένωσης. Ευχαριστούμε αγαπητέ συνάδελφε. Και τώρα εκ μέρους της ομάδας ID ο κύριος Φάντεντρισε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, τα τελευταία χρόνια έχουμε ε, πλημμυρίσει από κύματα προσφύγων, αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή. Ο πληθυσμό τη Αφρική θα μεγαλώσει δισεκατομμύρια ε, αυτών τον αιώνα μόνο και εκατομμύρια από αυτού θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να διαχειριστούμε σωστά τα σύνορά μα. Όχι γιατί μισούμε όσου βρίσκονται εκτό, αλλά γιατί αγαπούμε αυτού που ήδη ζουν εντό των σύνορων. Οι, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, χρησιμοποιούν ως εργαλείο τους ε, τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες. Θέλουν να γίνουν Ε, να γίνουν ε, ένα μέσο για να προωθήσουμε την ε, έλλειψη ελέγχου που επικρατεί εκτός των συνόρων μας. Γίνονται εργαλείο λοιπόν τα ανθρώπινα δικαιώματα για να ξεκινήσει ένα άνοιγμα των συνόρων και να υπάρξει εισβολή νέων πληθυσμών. Θα πρέπει το πρόβλημα να λυθεί στο επίπεδο των συνόρων μας και στη φύλαξή τους και να ε, μην επιτρέψουμε σε όποιον είναι οικονομικό μετανάστη επειδή απλώς το θέλει να ε, έρθει στην ε, Ευρώπη. Όσοι δεν έχουν δικαίωμα να φτάσουν εδώ θα πρέπει να παραμένουν στη χώρα τους. Ευχαριστούμε κυρία Φαντεντρίσε και τώρα εκ μέρους των Πρασίνων ο κύριος, η κυρία Στρίκ για μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εάν μιλήσουμε για κοινά εξωτερικά σύνορα, πρέπει να μιλήσουμε και για κοινέ ευθύνε όχι μόνο για τον έλεγχο όσων έρχονται προ τα μέσα, αλλά και για το πώ μεταχειριζόμαστε τον κόσμο. Πρέπει να έχουν μια ε, κανονική διαδικασία ασύλου στη διάθεσή του. Πρέπει επίση να του φερόμαστε με αξιοπρέπεια και να ε, ολοκληρώνονται οι διαδικασίε καταξής ε, των αιτήσεών του. Όμω σε πολλέ περιπτώσει στα σύνορα οι κανόνε δεν γεννητηρούνται. Οι αναπροωθήσεις είναι και οι αποθήσει είναι κάτι το καθημερινό στην Ευρώπη και θα υπάρξει απόφαση αύριο από το δικαστήριο του Στρασβούργου κατά τη Ισπανία. Υπάρχουν βίες ε, αποκρούσει και αποθήσει, ιδίω στα σύνορα τη Κροατία, ε, όπω έχουμε δει από πολλαπλέ μαρτυρίε και στοιχεία. Ε, την περασμένη εβδομάδα, σε επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε, σοκαριστήκαμε το γεγονό ότι όλοι που συμμετέχουν στη φυλακή των σύνορων, οι βίε πράξει και οι βίε αποκρούσει των μεταναστών είναι κάτι το καθημερινό. Και όμω τα διαψεύδει και τα αρνείται η κυβέρνηση τη χώρα. Αυτό δείχνει ότι η βία δεν θα σταματήσει, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να κάνει στραβά μάτια και να αντιδρά διαφορετικά. Ε, θα πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε πιστοί στι αξίε και τι αρχέ μα. Αλλά αυτό το δείξουμε αν κάνουμε κάτι για τι παραβιάσει των δικαιωμάτων στα σύνορα και φροντίσουμε να επιταχυνθεί και να ενταθεί η συμμόρφωση. Θα πρέπει να ε, μελετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ερευνήσει τι καταγγελίε και ε, τα παράπονα. Και θα πρέπει επίσης αυτές οι αξιολογήσεις να είναι μέρος το πώς λειτουργούν ε, ε, τα σύνορα και φύλαξη του χώρου Σέγγεν. Θα πρέπει να δούμε ότι τα χρήματα που παίρνει η Κροατία δεν πηγαίνουν στη φύλαξη των σύνορων, αλλά για τη φύλαξη των ε, περιοχών όπου γίνονται οι επαναπροωθήσεις. αυτή δεν επιτρέπεται, αυτοί που θέλουν να μελετήσουν τις επαναπροωθήσεις ή τις αποκρούσεις δεν επιτρέπεται να φτάσουν στην πράσινη ζώνη όπου αποκρούνται οι μετανάστες. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις παραβιάσεις, τις κατάφορες ε, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα. Τι συγκεκριμένα βήματα θα λάβει για να διακοπεί Συνάδελφοι, σα παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο ομιλία σα. Εκ μέρου των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριο Μπρουτζίνσκι. Για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Το να καταπολεμήσουμε τα γενεσιουργά της τη μετανάστευση είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία τη διαχείριση τη μετανάστευση. Και ποια είναι τα γενεσιουργά αίτια. Πρώτα απ' όλα, η αστάθεια, ο πόλεμος των χωρών που βρίσκονται γεωγραφικά κοντά και η έλλειψη ε, ε ανάληψης ευθυνών. Καλώς ήρθατε στον 21ο αιώνα. αυτό που είπαν οι Γερμανοί, το Herzlich Willkommen, το καλώ ήρθατε, δεν ισχύει. Ε, οι πρόσφυγε δεν έφτασαν εκεί που έπρεπε γιατί του πήραν τη θέση οι οικονομικοί μετανάστες. Ω τώρα λοιπόν η επίδραση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι γειτονικέ χώρε και τα όσα κατάφερε δεν ήταν αρκετά. Οι πραγματικές ε, απειλέ δεν περιορίστηκαν και αυτό μπορεί να δημιουργήσει να, και άλλη μεταναστευτική κρίση με την οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε στο μέλλον. Ε, άρα, πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Θα πρέπει να έχουμε ε, στοχευμένα μέτρα και τα κράτη-μέλη να δείξουν και καλή. Ευχαριστώ, αλλά αν συνάδελφοι συνεχίσετε να ξεπερνάτε το χρόνο αγόρευσή σα, θα ανάγκωσουμε να σα κόβω ε, το λόγο. Για, μην αναγκάσετε να το κάνω. Εκ μέρου τη ΓΚΟΕ, η κυρία παρακαλώ. Η συνοριακή πολιτική ε, είναι ευρωπαϊκή πολιτική και όχι εθνική. Είναι αλήθεια επίση ότι η πολιτική ασύλου και μετανάστευση χρειάζεται ευρωπαϊκή λύση. Μπορώ να καταλάβω ότι η Κροατία λόγω της ε, καταστροφικής κατάστασης που επικρατεί στα ελληνικά ε, hot spot, όμως διακινδυνεύει να γίνει η ίδια ολόκληρη ένα hot spot. Όμως αυτό δεν δίνει το δικαίωμα στην κροατική αστυνομία να βασανίζει, να ε, χτυπά πρόσφυγες με μασκοφόρους, να τους επιστρέφει στη Βοσνία, να τους κλέβει τα κινητά τους τηλέφωνα, τα χρήματά τους, να τους αφήνει ακόμη και όταν χρειάζονται βοήθεια, ιατρική περίθαλψη. Εν, το να κλείνουμε τα μάτια σε έναν τέτοιον σαδισμό δεν είναι ευρωπαϊκή λύση. Υπάρχουν ε, κανόνες όπως είναι η Σύμβαση για την Εξάλληψη των Βασανιστήριων για παράδειγμα που ισχύουν και για την Κροατία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν παντού και φυσικά και στα σύνορα. Ευχαριστούμε ο κύριος Παπαδάκης για ένα λεπτό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, συνεχίζοντας από τον ΣΥΡΙΖΑ την ευρωενωσιακή πολιτική καταστολής, χτίζει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου φυλακές στα ελληνικά νησιά, όπου με βάση και τη γερμανική πρόταση για το Δουβλίνο θα συνεχίζει να εγκλωβίζεται ο κύριος όγκος των ετούντων άσυλο. Η πλειοψηφία απέλαση, ελάχιστη άσυλο και ακόμα πιο λίγοι θα πηγαίνουν τελικά σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης. το τι πραγματικά ετοιμάζεται φανερώνεται από την διεύθυνση επιστροφών που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή μια φάμπρικα απελάσεων για να γυρίζουν οι πρόσφυγες πίσω στην κόλαση του υπεραλιστικού πολέμου που ευρωπαϊκή ένωση ηπα νατο κυβερνήσεις φουντώνουν έχοντας τεράστιες ευθύνες να πάρθει πίσω η υπογραφή της ελλάδας από τη συμφωνία ευρωπαϊκής ένωσης τουρκίας και από τον κανονισμό του δουβλίνου να καταδικαστεί η πολιτική των δολοφονικών πλωτών φραγμάτων παγίδων της εμπλοκής και χρηματοδότησης ΜΚΟ, της ανοχής στη δράση ακροδεξιών ομάδων που πυροδοτεί εντάσεις στα νησιά σε μια ούτως ή άλλως πολύ δύσκολη κατάσταση για νησιώτες και πρόσφυγες να κλείσουν τα hot spot με κέντρα φιλοξενίας στην ενδοχώρα για μετάβαση στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Και τώρα ο κύριος Σόκολ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πραγματικά απίστευτο το γεγονός ότι για άλλη μια φορά συζητούμε ψευδείς ειδήσει σχετικά με την, ε, με την δίθεν κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ε, από την κροατική αστυνομία, με ευθύνη της κροατικής ε, αστυνομία. Είναι τελείως μονομερής η πληροφόρηση. Από οργανώσεις που υποτίθεται ότι υπεσπρίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά στην πραγματικότητα θέλουν, ε, στόχο, στόχο έχουν να αποτρέψουν την είσοδο της Κροατίας στο Σέγγεν. Ούτε καν ξέρουμε για ποιου ανθρώπου μιλάμε. Μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι έχουν πέντε και 6 φορέ προσπαθήσει να διασχίσουν παράνομα τα σύνορα και τι κάνουν αφού δεν τα κατάφεραν, κατηγορούν τις κροατικές αρχές. Όμως η Κροατία είναι αυτή που διαφυλάσσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταπολεμά την παράνομη μετανάστευση και διαφυλάσσει τα 300 χιλιόμετρα εξωτερικών της ε, ε, συνόρων και πέρσι μόνο σταμάτησε χιλιάδε ανθρώπου που προσπαθούσαν να εισέλθουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, συνέλαβε 959 λαθροδιακινητέ ανθρώπων. Αυτό είναι αυτό που ενοχλεί σε, σε ό,τι αφορά τη στάση τη ε, ε, Κροατίας. Δέχεστε από την κυρία Έρνστ μια μπλε κάρτα. Έχετε το λόγο. Ναι, εκπλήσωμε υπάρχουν ε, άπειρες αποδείξεις ότι υπάρχουν μαζικές επαναπροωθήσεις και αποθήσεις στα κροατικά σύνορα και ότι σχεδόν όλοι οι μετανάστες που έχουν πληγεί από αυτό ε, το έχουν, έχουν δεχτεί μια τέτοια μεταχείριση τρεις και τέσσερις φορές χωρίς να έχουν ε, ποτέ αποκτήσει πρόσβαση στο δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα ασύλου. Τα έχετε ακούσει ποτέ αυτά. Δεν έχετε ακούσει τις κατηγορίες από μετανάστες και πρόσφυγες ότι έχουν ε, έχει ασκηθεί βία εναντίον του. Δεν τα έχετε ακούσει αυτά. Θα αναγνωρίσετε ποτέ την ε, πραγματικότητα. Είστε διατεθειμένος. Ε, Παρακαλώ. Ναι, στη ζωή μου έχω ακούσει πάρα πολλά ψέματα. Όμως το να επαναλάβει κανεί χίλιε φορέ ένα ψέμα δεν, δεν το καθιστά πραγματικότητα και αλήθεια. Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να αξιοποιήσουν και να εκμεταλλευτούν τι τις του συστήματο ασύλου και προσπαθούν να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή επικράτεια χωρί καθόλου να προέρχονται ή να κατάγονται από εμπόλεμε περιοχέ. Υπάρχουν και άνθρωποι που έρχονται από χώρε που δεν έχουν καθόλου πόλεμο. Φυσικά αυτοί οι άνθρωποι λένε ψέματα και αυτά τα διαδίδουν δυστυχώ και οι μη κυβερνητικέ ε, οργανώσει. Εγώ δεν μπορώ να τα πιστέψω Αυτά ίσως εσείς μπορείτε να τα πιστέψετε. Ευχαριστούμε και τώρα κυρία Σάντους για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την φρικτή κατάσταση των προσφύγων και μεταναστών σε διάφορα σημεία του κόσμου. Όμως πάνω από όλα στις πύλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως δείχνει το σύνορο μεταξύ Κροατίας και Βοσνία Αρζεγοβίνης, που η Κροατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχουμε δει και είχαμε αποδείξεις, ε, μαρτυρίες ε, δραματικές για την απάνθρωπη μεταχείριση των προσφύγων από την Κροατική αστυνομία κατά την απόθυση ανθρώπων που δεν είχαν καμία δυνατότητα να φτάσουν κανονικά στην επικρατεία τη χώρα και να αποβάλουν οποιαδήποτε αίτηση. Πολλέ φορέ έχασαν τη ζωή του στην προσπάθειά του να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει εδώ την ευαισθησία τη. Ε, θα μπορούσα να δείξω και σοκαριστικέ φωτογραφίε ε, με το τέλο τη παρέμβασή μου, αν θέλετε να έχετε απτέ αποδείξει. Στην Κροατία λοιπόν μιλήσαμε με πολλού πρόσφυγε και μετανάστε, νέου που ακόμη δεν έχουν φτάσει τα 18 και ε, δεν είχαν την, καμία δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε διαδικασία ασύλου και βρίσκονται ε, εκτός ε, τα μέλη της οικογένειάς τους προσπαθώντας να ε, ασκήσουν αυτό το περιβόητο δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης. Πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτά τα άτομα να βγουν από το λίμπο στο οποίο έχουν ξαφνικά βρεθεί και στο απόλυτο κενό. Θα πρέπει να υπάρξουν νόμιμοι διάβλοι και ταχείες διαδικασίες που με τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις να, ή τις φοιτητικές και θεωρήσεις να επιτρέψουν την οικογενειακή επανένωση. Δεν, μπορούν να, δεν μπορούμε να παραμείνουμε ούτε στη σιωπή ούτε στην αδιαφορία. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφε Σάντου, υπάρχουν ε, ερωτήματα με τη γαλάζια κάρτα. Τα δέχεστε, ε, κυρία Κλάβα, πρώτα απ' όλα. Διότι έχω πει ότι θα δέχομαι μία γαλάζια κάρτα ω τώρα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να δίνω το δικαίωμα τη γαλάζια κάρτα στον συνάδελφο που πρόλαβε Παρακαλώ να δείξετε κατανόηση. Δέχεστε κυρία Σάντο τη γαλάζια κάρτα τη κυρία Γκλάβακ. Παρακαλώ. Κυρία Γκλάβακ. Συνάδελφε, θέλω απλώ να ρωτήσω το εξή. Δυστυχώ, Η Κροατία έχει πολύ κακές μνήμες από την σερβική εισβολή ε, και είχαμε ε, εκατοντάδε, δεκάδε χιλιάδε μεταναστέ. Δεν καταλαβαίνετε. Εγώ ζω στην Κροατία. Η Κροατία κάνει ό,τι μπορεί ώστε η πρόσβαση στα κροατικά σύνορα να γίνεται ε, νομίμω και βάσει όλων των κανόνων και του διεθνού δικαίου. Και βάσει αυτού του διεθνού κοινέου δεν έχουμε τείχου και δεν έχουμε φράγματα σε σχέση με, με άλλε χώρε. Κοιτάξτε, προστασία των σύνορων δεν σημαίνει παραβίαση του διεθνού δικαίου οι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εάν η Κροατία θέλει να προστατεύει τα σύνορά τη, ε, χωρί να παραβιάζει το διεθνέ δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε γιατί ακόμη δεν εφαρμόζει το μηχανισμό παρακολούθηση όσων συμβαίνουν. Γιατί και γιατί τώρα χρειάζεται ένα ολόκληρο κοινοβούλιο να ζητήσει έρευνα για να μπορέσουμε να διαλευκάνουμε το τι πραγματικά συμβαίνει. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, και τώρα η κυρία Παγκαουρφουντούα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επίτροπε Ντελή, εάν κατάλαβα καλά, είπατε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν ισχύει αυτό. Δεν κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γνωρίζουμε ότι δεν αποδίδει ο κανονισμός του Δουβλίνου. Ε, παρ' όλα αυτά δηλαδή, το έχει μπλοκάρει το Συμβούλιο, δεν έχουμε κάποια πολιτική ασύλου, τόσο ώστε να σταματήσουμε αυτή την τραγωδία. Δεν κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, είπατε ότι ήδη έχουμε πετύχει πολλά. Τι, ότι η Μόρια, η Σάμος, η Χίος είναι μια κόλαση και η Λιβύη που είπατε ότι εκεί βοηθούμε για να ελαφρώσει η κατάσταση. Ε, όχι, δεν θα, αν δεν κάνουμε το πιο σημαντικό, δεν θα τους ελαφρύνουμε τη θέση. Θα πρέπει να κηρύξουμε την Λιβύη μια ασφαλή χώρα. Να, τι είναι στο χέρι μας. Πότε πρόκειται να κάνουμε ό,τι πραγματικά μπορούμε, κυρία Ντέλη, τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι λόγια. Εμείς λέμε ό,τι να είναι, γιατί λέμε ότι ε, θα αυξήσουμε κατά 40 το προσωπικό στα σύνορα, ας πούμε, ενώ γίνονται εκεί φοβερά πράγματα. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Μπαρντελά για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, το, το, το περίφημο προσφυγικό ξεκίνησε το 2015 τι κρίση είναι αυτή. Έχουμε όλους αυτούς ως ρε μπαίνουν στην Ευρώπη και όλοι αυτοί μας έχουν πνίξει. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο σε δύο χρόνια διπλασιάστηκαν οι ροές. Φτάσαμε στα 70.000 νέους ε, στο 19 στην ε, Σάμο. Έχουμε περισσότερους από όσο είναι οι κάτοικοι. Τι γίνεται με το σύνορο προς την Τουρκία, τι γίνεται με τον Εύρο όσα γίνονται εκεί δείχνουν πόσο η Frontex δεν καταφέρνει τίποτα και πόσο δεν ωφελεί η συμφωνία του 16 με την Τουρκία. Τα λέμε και τα ξαναλέμε ε, το με τι προϋποθέσεις ζουν, αλλά δεν κάνουμε τίποτα για τις αιτίες του προβλήματος. Οι υπεύθυνοι είναι αυτοί που με τις πράξεις τους και με τους λόγους τους ε, τους έχουν οδηγήσει να έρχονται στην Ευρώπη τους ανθρώπους. Πρόκειται για ένα δράμα. Χρειάζεται μια ανθρωπιστική αποτροπή, τέτοια πολιτική. Και αυτό να γίνεται ε, στα σύνορα και στις χώρες τους. Θα πρέπει να το πούμε και στην Τουρκία. Ε, τα πάει καλά η Ελλάδα να την βοηθήσουμε. Να μην τους ματιώσουμε τις προσπάθειες. Μα είναι δυνατόν κάποιος να μπορεί να φύγει αν διώκεται από τη χώρα του. Αλλά αυτό όμως να μην αναστατώνει τη ζωή ε, κάποιων σε άλλες χώρες που τους υποδέχονται. Σα Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα δίνει τον λόγο στον κύριο Μάρκαρτ για ένα μισή Ευχαριστώ πολύ. Εγώ μεγάλωσα στην Ευρώπη. Και καθώς μεγάλωνα, θεωρούσα πάντοτε ότι η παρεμβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κρατική ευθερεσία, οι ανθρωπιστικές κρίσεις είναι πράγματα που συμβαίνουν αλλού στον κόσμο, όχι σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά πήγα σε αποστολές ε, διάσωσης στη Μεσόγειο και τελικά διαπίστωσα ότι τελικά ενισχύονται περισσότερο οι Ισλαμικές πολιτοφιλικές από ότι οι οργανώσεις που προσπαθούν να διασώσουν ανθρώπους. Στην, ε, στην, ε, στην ε, Σάμο μίλησα με ανθρώπους από τη Σύρο οι οποίοι μου λέγανε γιατί οι ίδιοι οι ευρωπαϊκές αρχές μας, διαχειρίζονται, μας μεταχειρίζονται σαν ζώα. Στην Βοσνία Ερζεγοβίνη συμβαίνει το ίδιο. Το τι συμβαίνει στο, στην, στα εξωτερικά σύνορα νομίζω ότι δεν συνάδουν με την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας. Εγώ Είμαι, είμαι, πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως νομίζω ότι δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτό που πραγματικά θέλουμε να είμαστε. Αν η Κομισιόν είναι σοβαρή σε όσα λέει, πρέπει να δείξει στην Κροατία ότι ε, πρέπει να επιτραπεί ένας ανεξάρτητος μηχανισμός αξιολόγησης της στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα συνεργαστούμε μαζί με Ευρωπαίους αξιωματούχους ε, το τι συμβαίνει στα εξωτερικά σύνορα, ακριβώς γιατί θεωρώ ότι και η Κροατία δεν υπάρχει λόγος να κρύβει τα όσα συμβαίνουν. Εσείς όμως αρνείστε να δημιουργηθεί ένας τέτοιος ε, μηχανισμός. Έχετε μια μπλε κάρτα. Την δέχεστε. Έχετε το λόγο. Συνάδελφε, το μικρόφωνο σας λέει ο πρόεδρος. Κύριε Μάρκαρντ, εγώ ήμουν πρόσφυγας στην διάρκεια του πολέμου της πρώην Ιουγκοσλαβίας και έχω εργαστεί επίσης με δικηγόρους για την κατάσταση προσφύγων. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να διαπιστώσει κανείς αν υπάρχει αστυνομική αυθαιρεσία. Αυτό που λέτε είναι ψέμα, είναι ψευδές, μην το κάνετε, μην χρησιμοποιείτε τους πραγματικούς ετούντες άσυλο ε, για να διασπείρετε αυτά τα ψεύδη, διότι στην πραγματικότητα βλάπτετε τους πραγματικούς πρόσφυγες, συγκαλύπτετε τις ανθρώπινες τραγωδίες που πράγματι υπάρχουν, κατηγορώντας την κατηγορία. 100.000 Κροάτες ζουν στην Βοσνία Ερζαγοβίνη. Τους, έχει, τους δώσαμε κροατικά διαβατήρια στη διάρκεια του πολέμου και τους προστατεύουμε και αυτούς. Συνάδελφε Μάρκαρτ, μπορείτε να απαντήσετε. Ναι, κάτι είπα για αυτό το θέμα, όμως αναρωτιέμαι πάντοτε τι σημαίνει όταν εσείς κατηγορείτε εκείνους που κάνουν έρευνες, κρατικά ε, ΜΜΕ για παράδειγμα γερμανικά, που έχουν βίντεο από αποθήσεις βίες και εσείς λέτε ότι είναι fake news. Τι αντίληψη για την ελευθερία του τύπου είναι αυτή. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τι σημαίνει να χρειαστεί να γίνω πρόσφυγα. Όμω, μια και λέτε ότι εσεί ήσασταν πρόσφυγο, ίσω θα ήταν μια καλή ευκαιρία να μιλήσετε με του ανθρώπου που βασανίστηκαν, που του χτύπησαν οι αστυνομικέ δυνάμει, με αυτού του ίδιου ανθρώπου, για να δείτε ποια ακριβώ είναι η κατάσταση επιτόπου. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγο στον κύριο Φράγκο για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε απευθύνομαι στους έλληνες που μας κοιτούν από τις τηλεοράσεις στους υπολογιστές και τα κινητά τους απευθύνομαι στους κατοίκους της Σάμου, της Μυτιλίνης, των διαβατών και της υπόλοιπης ελλάδας που έχουν δει τον τόπο τους να μετατρέπεται σε ένα απέραντο χαλιφάτο. είναι πια δεδομένο πως η ευρωπαϊκή ένωση εξυπηρετεί τα συμφέροντα ατόμων όπως του σόρος που μέσω των ΜΚΟ και των μουσουλμάνων αποσκοπούν στο να εξαλειφθεί ο χριστιανισμός και να γεμίσει με τζαμί η ευρώπη. εμείς πρέπει να τιμήσουμε τις αξίες και τις παραδόσεις που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας. είναι ντροπή η ευρωπαϊκή ένωση να χρησιμοποιεί τα χρήματα του ευρωπαίου φορολογούμενου για να παρέχει δωρεάν διαμονή και διατροφή στους λαθρομετανάστες τη στιγμή που υπάρχουν έλληνες που λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν φτάσει να κοιμούνται στα αυτοκίνητά τους. εμείς η ελληνική λύση απαιτούμε μια ευρωπαϊκή ένωση χριστιανική που θα έχει στον πυρήνα της τον ιερό θεσμό της οικογένειας και όχι μια ευρώπη πολυπολιτισμική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο λόγος στον κύριο Αρβανίτη για να λεπτό. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν έχουμε χάσει κάποια από κάποιες ομάδες έχουν χάσει την ουσία της κουβέντας. Σήμερα μιλάμε για τα ευρωπαϊκά σύνορα. Και πρέπει να τονίσουμε ότι την αξία του πρόσφυγα και την αξία του μετανάστη είναι άλλες έννοιες. Φεύγουν από τη δικιά τους κόλαση λοιπόν από τον πόλεμο και εδώ στην Ευρώπη βιώνουν την ευρωπαϊκή κόλαση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και μάλιστα με νόμιμη κρατική βία. Τη βία των αστυνομικών, των συνοφυλάκων, την κρατική καταστολή. Στη Σερβία, στη Βοσνία, Ζεγοβίνη, στην Κροατία, στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία. Γίνονται καθημερινά καταγεγραμμένα εκατοντάδε περιστατικά βίαιων αποθήσεων. Έχουμε μαρτυρίε, είμαστε εμεί οι ίδιοι αυτόπτε μάρτυρε. Πήγανε εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου. Και όταν δείχνουμε τις εικόνες σοσιαλιστές πράσινοι αριστεροί βουλευτές ευρωβουλευτές των κατασπαραγμένων από σκυλιά της αστυνομίας ανθρώπων οι δύο υπουργοί της κροατίας λένε ότι αυτό είναι fake news και το ακούω και εδώ αυτό είναι προσβολή για τους βουλευτές αυτό είναι προσβολή για τις πολιτικές ομάδες που κάνετε. να ακούτε να ακούτε επιτέλους είναι ακροδεξιά ρητορική σας έχει μείνει μόνο το id και η ακροδεξιά. Και θέλω να σα πω ότι στην Ελλάδα τοποθετούν φλωτά φράγματα. Στα ελληνοτουρκικά σύνορα εκατοντάδε πεθαίνουν από πνιγμό και κρύο και θέλω να κάνω μια ερώτηση τελευταία απλώ να μα πει η ευρώπη τελικά την πρότασή σα όχι έκθεση ιδεών. τι πρόταση έχετε να μα πείτε. Thank you, sir. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Πονσατή Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Δεν μπορούμε να βλέπουμε ως ένα θέμα εξωτερικής ε, πολιτικής, ε, εξωτερικό που δεν μας αφορά τους πρόσφυγες. Γιατί πολλούς από εμά μας έχει καθορίσει γενιές Ευρωπαίων, όπως στη χώρα μου όσοι ξέφυγαν από ε, την φρίκη του φασιστικού καθεστώτος του Φράγκο πριν από 81 χρόνια σώθηκαν χάρη στο καθεστώς του πρόσφυγα και υπάρχουν παιδιά και εγγόνια προσφύγων που ζουν σε αυτό το κοινοβούλιο που ε, ξέρουμε ότι οι παππούδε μα, μπορεί να μην είμαστε εμεί και προπαππούδε μελλοντικών προσφύγων. Όμω το να ειναι κανεις κανεί πρόσφυγα πηγαίνει χέρι-χέρι με το να είναι κανεί και ένα ε, καλό οικοδεσπότη. Στην Ευρώπη θα πρέπει να φτιάξουμε ένα ασφαλή λιμένα για πρόσφυγες θα πρέπει ο καθένας που προσπαθεί να δραπετεύσει από εμπόλεμες περιοχές είτε είναι ε, πόλεμος οικονομικός είτε πόλεμος με πραγματικά όπλα να μπορεί εδώ να βρει ένα ασφαλή λιμένα, ένα ασφαλές καταφύγιο. Όχι ε, να υπάρξει απεικιοκρατία ξανά αλλά ε, ειρήνη και δικαιοσύνη στον κόσμο. Ευχαριστούμε. Ντυπώ για ένα λεπτό. Συνάδελφοι, στην προηγούμενη Ολομέλεια συζητήσαμε για την κατάσταση στα ελληνικά νησιά. Σήμερα συζητάμε και για τα εξωτερικά σύνορα στην Κροατία. Και στι δύο περιπτώσει η πολιτική ασυλίου και μετανάστευση μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν είναι ε, σύμφωνη με το ε, διεθνέ και το ε, ευρωπαϊκό δίκαιο και αν τηρεί ανθρωπιστικά πρότυπα. Όμω χρειάζεται να υπάρχουν και αυστηρέ κυρώσει. ο ε, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κροατία, καθώς και για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξωτερικά σύνορα, πρέπει να υπάρχει σαφής η δήλωση ότι περιμένουμε από εσά να διαφυλάτε τα σύνορά μας, αλλά δεν θα σας αφήσουμε και μόνους σας. Γι' αυτό και ζητούμε από την ε, Κομισιόν και το Συμβούλιο. Κοιτάζοντας τους αυξανόμενους ε, αριθμούς των μεταναστευτικών ροών, την αστάθεια στη γειτονία, πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την περίοδο αυτή ε, για να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα για το μέλλον, τότε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Ένα λεπτό, Λόπες Αγγιλάρ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Δεν έχουν ιατρική κάλυψη, υποφέρουν, δεν έχουν νομικές συμβουλές, δεν ενημερώνονται. Αυτό είναι κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου. Τι γίνεται με την οδηγία του 13 για το άσυλο. Θα πρέπει, υποχρεούται όπου χρειάζεται να παρέμβεται. Εκεί που έχουμε τέτοιου είδους επαναπροωθήσεις, έχουμε καταπάτηση του τετάρτου πρωτοκόλου ε, της Σύμβασης των Δικαιωμάτων και του χάρτη. Ε, δεσμεύει όλα τα κρατη όπου και να γίνεται ένα συμβάν. Άρα θα πρέπει να ξεκινήσετε διαδικασία παραβάση και να ε, υπάρχει βοήθεια από τα ευρωπαϊκά ταμεία, από όλα τα κράτη-μέλη, αλλά και ε, να βοηθάει και το σχετικό ταμείο ασύλου. Ε, θα πρέπει να το εξασφαλίσετε, να υπάρχει προσβασιμότητα, να μην υπάρχει καμία επαναπρόθεση προς χώρες όπως η Λιβύη. Θα πρέπει να ανοίξετε νόμιμους ασφαλείς διάβλους και έτσι να μην εκτίθενται ανθρώπινες ζωές, ανθρώπινες ζωές ακριβώς όπως ζήτησε στην προηγούμενη θητεία το Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το καθήκον σας για αυτή τη θητεία κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει μια μπλε κάρτα από την κυρία Σόντροβα κύριε συνάδελφε. Την δέχεστε. Μάλιστα έχετε το λόγο. Μικάλα. Ευχαριστώ πολύ αυτό που συζητούμε σήμερα σχετίζεται με το πόσο ανοιχτή πρέπει να είμαστε με την ανθρωπιστική υποδοχή χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών. Εγώ συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελέσει έναν ασφαλή λιμένα για όσους ανθρώπους χρειάζονται βοήθεια. Όμως, τον Σοσιαλιστή Υπουργό Εσωτερικών της Τσεχίας θέλω να τον καλέσω να να τον καλέσω, να του υπενθυμίσω μάλλον ότι του ζήτησα να, έρθει να φέρει 50 ασυνόδευτα ε, παιδιά από τη Συρία. Δεν κατονόμασα καμία χώρα και κανένα κόμμα. Όποιος βρίσκεται εδώ δεσμεύεται από τη συνδίκη τη Λισαβόνα από τον χάρτη για τα θεμελιώδη δικαιώματα, το ανθρωπιστικό δίκαιο, δεσμεύει όλες τις χώρες και την ειδική σας. Δεν υπάρχει διέξοδος από αυτή την ε, υποχρέωση. Δεσμευόμαστε 100% σε σχέση με ε, το άσυλο. Σήμερα εγκρίναμε το φάντο ακριβώς για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφαλή λειτουργία της ελεύθερης διακίνησης προσώπων. Αλλά σε όλα τα κράτη-μέλη ε, την χάνει προστασία και που επικαλείται το ανθρωπιστικό δίκαιο. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα η κυρία Γιώβεβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ακούμε αναφορές σχετικά με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, προσφύγων και μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων και των Κροατικών. Και μιας και ε, είναι στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου φέτο η Κροατία, έχουμε και εκπρόσωπο. Εσεί λέτε ότι δεν υπάρχουν αποδείξει για όλα αυτά. Θα σα πω εγώ το εξή. Τον προηγούμενο μήνα, μια ομάδα μη κυβερνητικών οργανώσεων εξε, εξέδωσε μια έκθεση που αποδεικνύει ότι οι κροατικέ αρχέ χτυπά με λοστού του ανθρώπου αυτού, με ε, όπλα και του αποθεί στη Βοσνία ακόμη και οι αρχές του ΟΗΕ, ακόμη και ορισμένοι Κροάτες αστυνομικοί έχουν βγει και έχουν κάνει καταγγελίες. Και τι απάντησαν οι κροατικές αρχές, ότι αυτά τα κάνουν για να μπορέσουν να, να ικανοποιήσουν τα κριτήρια του Σέγγεν. Να σας πω κάτι, Μπορεί να πάω κι εγώ. Να το αποφασίσω και να πάω εγώ. Να πάρω τη φωτογραφική μου μηχανή και να πάω να σα δείξω εγώ η ίδια τι συμβαίνει εκεί. Ευχαριστούμε. Υπάρχει γαλάζια κάρτα από το, για εσά από την κυρία Ρέσλερ. Τη δέχεστε, Ρέσλερ. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, όσοι θέλουν ε, να έχουν διεθνή προστασία μπορούν να την ετηθούν. Και αυτό βάσει ε, ε, των διαδικασιών που μπορούν να εφαρμοστούν στα επίσημα σημεία διόδου και με τα ταξιδιωτικά έγγραφα που θα πρέπει να κατέχουν. Όμως υπάρχουν πολλά επεισόδια, όπως είπατε, που ίσως Ε, να έχουν να κάνουν και με τον αριθμό, ασύλ, αριθμό αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή. Όσοι περνούν τα σύνορα δεν θέλουν να περάσουν από τα επίσημα ε, σημεία ελέγχου στη σύνορα, στα σύνορα, στη συνορφυλακή. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, δεν μιλούσα για τις ελάχιστες απαιτήσει και για τις διαδικασίες αίτησης ασύλου. Εδώ μιλάω για τα εξωτερικά σύνορα της Κροατίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κροατία. Τώρα λέτε ότι όλα αυτά είναι ψεύδι. Τι να πω, ίσω ζούμε σε παράλληλου κόσμου. σω θα πρέπει να πάμε να πιούμε ένα καφέ και να κοιτάξουμε μαζί τι φωτογραφίε και τα βίντεο, μπα και σα πείσουμε. Αλλά έχω πάει η ίδια, η ίδια εκεί ω δημοσιογράφο. Θα πάω και ω πολιτικό. Και με μεγάλη μου χαρά και μακάρι να αποδειχθεί ότι έχετε ε, δίκιο εσεί και όχι εγώ. Αλλά μπορώ να σα φέρω και φωτογραφικό υλικό. Ευχαριστούμε ο κύριο Μπλάσκο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πραγματικά κρίμα που ε, ε χιλιάδε μετανάστε στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Εδώ θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να μπορέσουν να κοιτάξουν πώς θα διαχειριστούν αποτελεσματικά βάσει των ε, ε, βασικών προϋποθέσεων το θέμα της μετανάστευσης. Βεβαίως δεν μπορεί να έρχονται μετανάστες εδώ μόνο με σκοπό μια καλύτερη ανετότερη ζωή ε, και για να εκμεταλλευτούν τα κοινωνικά ωφελήματα του ευρωπαϊκού συστήματος. Θα πρέπει να μην ε, χάνουν δικαιώματα οι δικοί μας ε, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι και αυτά να δίδονται στους μετανάστες. Υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν πληρώσει εισφορές όλη τους τη ζωή, έχουν εργαστεί όλη τους τη ζωή και δεν είναι εξίσου προστατευμένοι όπως οι μετανάστες. Εδώ λοιπόν, εάν δεν καταλαβαίνετε ότι αυτά συμβαίνουν λόγω της ε, πολιτικής σας που δεν έχει καμία λογική, τότε γεμίζετε με μετανάστες και πρόσφυγες στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Μπέζελάγκερ για ένα λεπτό. Πριν από δύο εβδομάδε είχαμε συζητήσει την κατάσταση στα ελληνικά νησιά και βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στην πράξη από τότε που μιλήσαμε γι' αυτό. Ε, η απάνταση είναι ότι τα πράγματα έχουν επιδονωθεί. Από το ευρωπαϊκό επίπεδο δεν καταφέραμε να κάνουμε τίποτα για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Ναι, χρήμα στείλαμε για να δημιουργηθεί ένα πλωτό φράγμα και να μπορέσουν να ε, μείνουν εκτός όσοι κάνουν αιτήσει ασύλου. Τώρα διαμαρτύρονται και οι ντόπιοι και οι πρόσφυγες για όσα προγραμματίζονται. Σταματήσουμε λοιπόν το παιχνίδι επίληψη ευθυνών μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπή και από τι δύο πλευρέ α κοιτάξουμε να αναλυφθεί δράση για να βελτιωθεί κατάσταση στην πράξη. Δηλαδή να ξεκινήσουν οι μηχανισμοί προστασία των πολιτών και να λειτουργούν ε, να ενεργοποιηθούν τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Δηλαδή, οι ανήλικοι και οι συνόδευτοι ανήλικοι που χρειάζονται τη βοήθειά μα τόπου να ε, προσκληθούν και να έρθουν σήμερα. Να δράσουμε σήμερα και όχι μεθαύριο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε. Και τώρα ο λόγο στον κύριο Τζαμπάσκε για ένα λεπτό. Όλια, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούω να επικρίνετε την Κροατία. Αυτό είναι αβάσιμο δεν μπορείτε να κατηγορείτε Κροατία, Ελλάδα, Βουλγαρία. Γιατί οι δικές μας χώρες σας προστατεύουν από τους ε, μουσουλμάνους, τους τζιχαντιστές, τους τρομοκρατίες. Εμείς φρενάρουμε εκείνους που ήρθαν για να εισβάλλουν στις ευρωπαϊκές πόλεις. Σε κάθε χώρα θα πρέπει να προστατεύσει τα σύνορά της. Δεν είναι δυνατόν ε, να ζητάτε να αφήσουν αυτές οι χώρες τον κόσμο ε, τους τρομοκράτε μέσα στα σύνορά του. Πρόκειται περί φαρισαϊσμού. Εσείς ε, λέτε ότι νοιάζεστε για αυτού του ανθρώπου. και ε, τότε σηκώστε το χέρι σας όσοι από εσά έχετε συμφωνήσει να έρθετε στη χώρα σας τζιχαντιστή, αυγανός τρομοκράτη, να έρθει στο σαλόνι σας με τα παιδιά σας να κάτσει. Περιμένω πώς και πώ να δω ποιο θα σηκώσει το χέρι του. Ε, δεν βλέπω και κανέναν, οπότε σταματήστε την υποκρισία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον ε, λόγο έχει κυρία Γουόλς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Απορώ που δεν σκόθηκε καμία μπλε κάρτα μετά από τον συνάδελφο. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι τεράστιες. Βλέπουμε έκρηξη στον αριθμό των ανθρώπων που αναζητούν μια καλύτερη ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μακριά από τη φτώχεια και τη βία και τις καταστροφές. Οι φρικτές συνθήκες σε οποιαδήποτε από τα στρατόπεδα, σε οποιαδήποτε από τι χώρε για τι οποίε μιλάμε, ε, σημαίνει ότι υπάρχει φοβερή πίεση από τους ανθρώπους που είναι ευάλωτοι και τους άλλους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνθήκες είναι αφόρητε και τα λόγια δεν κάνουν τίποτα. Δεν μπορεί να επομίζονται το βάρος λίγες χώρες. Χρειάζεται η βοήθεια της Ευρώπης θεωρώ πως το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι θύμα της ίδιας του της επιτυχίας. Πρέπει λοιπόν να επιδείξουμε μεγαλοψυχία και αλληλεγγύη για να στηρίξουμε και τα κράτη-μέλη μας τα οποία βλέπουν την μεγαλύτερη εισρωή. Έχει τελειώσει ο χρόνος μου. Θα πω ότι χρειάζεται μια ανθρωπιστική και στρατηγική λύση. Και τολμώ να πω, μια άμεση λύση είναι να γίνει αυτή η συζήτηση Ε, αλλά με λίγο περισσότερους βουλευτές από τους 40-50 που είναι εδώ μέσα. Σας ευχαριστώ. Φόλαθ ε, για ένα λεπτό τώρα. Δύο φορές έχω πάει εγώ προσωπικά να δω την ανθρωπιστική κατάσταση στα κροατικά σύνορα, η οποία εξακολουθεί να είναι δραματική. Ειδικά η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων οι άνθρωποι εκεί και οι πολιτικοί έχουν ε, πελαγώσει από την κατάσταση και αισθάνονται ότι τους πούλησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πανηγυρικοί όπως οι σημερινοί λόγοι δεν βοηθάνε. Και το να κρύβουμε το κεφάλι στην άμμο βλάπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ περισσότερο από τον Brexit γιατί καταστρέφει την Ευρωπαϊκή Ένωση φροντίστε επιγόντως για να ανακουφιστεί η ανθρωπιστική κατάσταση ειδικά των παιδιών που πρέπει να φύγουν από εκεί και να υπάρξει ανεξάρτητη παρακολούθηση των συμβάντων στα σύνορα. Επιτέλους, φτιάξτε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου χωρίς παράνομες αποθήσεις. Μόνο με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα θα υπάρξουν πραγματικές λύσεις. Αλλιώς θα χάσουμε την αξιοπιστία μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και... Να σας χαιρετήσω και εσάς και δίνω τον λόγο στην κυρία Σαρντώνε από το ID. Η... Μας λέτε ότι οι συνθήκες αυτές οφείλονται στην Ευρώπη και η Ευρώπη, η Ευρώπη είναι υπεύθυνη γιατί η Ευρώπη λέει υποδοχή με κάθε κόστος. Ε, προσπαθούν τώρα να επιζήσουν, τα έχετε φορτώσει στις χώρες της ε, περιφέρειας και οθούνται στο έγκλημα. Είναι υποκριτική η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ασχολείται με την κατάσταση των μεταναστών αλλά ασχολείστε μόνο με τις χώρες Μεσογείου. Γιατί δεν κάνετε τίποτα να σταματήσετε τις ε, αποβιβάσεις και να σταματήσετε κυρίως τις αναχωρήσεις Έχετε εδώ πέρα την Κάρολα Ρακέτε, τη Μίκη Ωμα. Ποιο το χρηματοδοτεί, Ποιο χρηματοδοτεί του ανθρώπου με τι βάρκε. Λοιπόν, τα έχουμε πει και με τον Ματέο Σαλβίνη. Τέρμα η παράνομη μετανάστευση και να σταματήσει επιτέλους αυτή η κατάσταση με την ανεξέλεγκτη υποδοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρουκ από το ΙΣΙΑΡ. Κυρίε και ε, αν ε, παρακολουθήσουμε τα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωση τη Ευρώπη, ε, θα νομίσουμε ότι η μεταναστευτική κρίση τελείωσε το 2016. Όμω εξακολουθεί να υφίσταται με δύο τρόπου. Ανθρωπιστικά στα εξωτερικά σύνορα και η μεταναστευτική κρίση εντό των ευρωπαϊκών σύνορων, εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2015 που ανοίξαμε τα σύνορα σε όλους. Στα ε, σύνορα οι περισσότεροι χαρακτηρίστηκαν ως πρόσφυγες παρόλο που οι περισσότεροι δεν ήταν πρόσφυγες αλλά οικονομικοί μετανάστες. Τώρα αντιμετωπίζουμε τα αποτέλεσματα εκείνης της πολιτικής. Ήταν μια σκόπιμη πολιτική που είχε στόχο να καλέσει εκατομμύρια μεταναστών στις, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τους ε, κάνει ε, Ευρωπαίους πολίτες, παρόλο που δεν είναι χριστιανοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται περισσότερου πόρου. Χρειάζεται καινούρια ιδεολογία και όχι τη μαρξιστική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο λόγο του κύριο Μέλο από το ΕΛΚ. Η μια Ευρώπη με ανοιχτέ πόρτε ε, είναι παράλογη. Ε, μόνο η αριστερά, ανεύθυνη αριστερά το υποστηρίζει. Δεν υπάρχει καμία χώρα του κόσμου που να έχει ανοιχτά σύνορα, που να επιτρέψει όλους να μπουν μέσα αρκεί να το θέλουν. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι διαφορετική. Θα πρέπει να σεβαστούμε αυτόν που θέλει να βελτιώσει τη συνθήκη ζωή του και έχουμε υποχρέωση να υποδεχθούμε με ανθρωπισμό του ανθρώπου. Όμω, θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί σε ό,τι αφορά τον έλεγχο τη εισόδου από τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να κάνουμε διάκριση. Άλλο οι πρόσφυγες, άλλο οι μετανάστες. Στους πρόσφυγες εφαρμόζονται διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικοί νόμοι από ότι αυτοί που εφαρμόζονται για τους μετανάστες. Αυτοί που θεωρούνται πρόσφυγε έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να σώσουν τη ζωή του και πρέπει να του υποδεχτούμε σύμφωνα με τι διεθνεί συνθήκε. Όμω, όποιο έρχεται απλώ για αναζήτηση εργασία ω μετανάστη, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με του εθνικού κανόνε τη κάθε χώρα και σύμφωνα με το χείρι τη επικουρικότητα. Κάθε χώρα γνωρίζει ποιου και πόσου μετανάστε χρειάζεται. Δεν είναι δυνατόν να συγχαίουμε αυτέ τι δύο κατηγορίε. Γιατί αλλιώ θα κινδυνεύσουν το, κοινωνικό, το εργασιακό και το δημοκρατικό μα σύστημα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ να σέβεστε το χρόνο που σας έχει δοθεί, ένα λεπτό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο συνάδελφο Νόιζερ ο λόγος για ένα λεπτό. Α, υπάρχει, υπάρχει μπλε κάρτα. Ε, Τη δέχεστε, δέχεστε την μπλε κάρτα, ναι. Αναφερθήκατε στη διαφορετική νομική βάση για πρόσφυγες και μετανάστες. Σωστό αυτό. Αλλά ένα ερώτημα προκύπτει. Οι μετανάστες έχουν παρόλα αυτά ανθρώπινα δικαιώματα ή δεν ισχύει αυτό και ισχύει μόνο για τους πρόσφυγες. Ε, εσείς πιστεύετε ότι